Μάλιστα. Λέω να αρχίσουμε. Γιατί φοβάμαι ότι η ανακοινώσει της Προεδρίας είναι πιο μακροσκελής τώρα που είμαστε στον τριμερή διάλογο. Λοιπόν, πρώτον η έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασης των όλων περασμένων συνεδριάσεων. Φαντάζομαι ότι εγκρίνονται. έγκριση των πρακτικών της 13ης Δεκεμβρίου 10-28 Φεβρουαρίου 7 Μαρτίου 16 Μαρτίου και 21 με 22 Μαρτίου έχουν διανεμηθεί φαντάζομαι ότι εγκρίνονται και αυτά και τώρα οι ανακοινώσεις της Προέδρου πρώτα και καλύτερα ανταλλαγή απόψεων με τον Επίτροπο Ρεν και την Προεδρία του Eurogroup τον κύριο Γιούνκερ που θα γίνει στη συνεδρίασή μας της 6ης Ιουνίου στο Στρασβούργο για την φάση στην οποία βρίσκεται ο τριμερής διάλογος για τα χρηματοπιστωτικούς ομίλους δεν έχουμε τίποτα πιο πρόσφατο για την λιανική Έχουμε τη θέση του Συμβουλίου από χθε. Έγινε μια παρουσίαση της Προεδρίας. Συζητήσαμε τη μέθοδο διαπραγμάτευσης και την ημέρηση διατάξη των επομένων τριμερών διαλόγων. Καμία απόφαση δεν ενημερώθηκε. Θα δούμε τι θα πούν οι διαπραγματεύσεις στο μέλλον. Για την οικονομική διακυβέρνηση governance Έχουμε συναντήσεις του τριμερούς διαλόγου στις 10 και 11 Μαΐ, είχαμε, Μαΐου. Και εκεί ξαναεξετάσαμε όλες τις εκθέσεις και αναφορές από την Προεδρία του Συμβουλίου. Υπάρχει ένα μακροκελές σημείο που θα διανεμηθεί στους συντονιστές και συντονίστριες. Και είμαι βέβαιο ότι δεν θέλετε να σας το διαβάσω τώρα φωναχτά αλλά όσοι δεν το λάβουν μπορούν να το ζητήσουν. Το ίδιο ισχύει και για τη συνεδρίαση του τριμερούς διαλόγου στις 17 Μαΐου όπου συζητήσαμε, συνεχίσαμε τη συζήτηση των οριζοντίων θεμάτων για τον οικονομικό διάλογο και τη σύνδεση με τους ε, στόχους 2020, τις μακροοικονομικές ανισορροπίες και ανισότητες και μετά και χθες έγινε ένας τριμερής διάλογος όπου η συζήτηση ήταν πιο λεπτομερής για τα οριζόντια θέματα και αρχίσαμε τη συζήτηση άρθρο προς άρθρο για την έκθεση κόλ. Θα γίνει το ίδιο και στον επόμενο τριμερή διάλογο την Τετάρτη το απόγευμα, 25 Μαΐου. Επίσης αυτή την εβδομάδα στις 5 σήμερα θα γίνει μια τεχνική συνάντηση μεταξύ γραμματείας και εκπροσώπων των θεσμικών οργάνων για την έκθεση ΦΕΑ. Και είναι ανοιχτή η συνάντηση αυτή σε όλους τους εισηγητές και τους κοιόδης τους. Επίσης συμφωνήσαμε ότι επειδή θα λείπω στην Ιρλανδία και όποτε άλλοτε χρειαστεί να λείπω για τον τριμερή διάλογο για την οικονομική διακυβέρνηση ο αντιπρόεδρος Σικούμνα θα με προσωπεί γιατί έχει ασχοληθεί ήδη με το θέμα και αυτή η πρόταση υποστηρίχθηκε ομόφωνα. Και τους υπόλοιπους αντιπροέδρους τους το ανακοίνωσα, δεν έθεσε κανείς αντίρρηση. Μερικοί μάλιστα το βρήκαν και καλό. Αυτό θα γίνει λοιπόν. Υπάρχει ένα μα αν θέλει οποιοδήποτε μπορεί να το ζητήσει, ούτως ή άλλως θα το στείλουμε στους συντονιστές. Στις ομάδες δηλαδή. Προφανώς και οι συγητές και οι συγητρίες καθώς και οι σκιώδεις. Ήταν πολύ πλήρης συνάντηση με περίπου 70 άτομα ή πρόσωπα. Πάμε τώρα σε δική μου έκθεση ο Θεέ μου. Μήπως δεν πρέπει να προεδρεύω ταυτόχρονα. Είναι η γραφή τη Ευρωπαϊκή Ένωση για την απόκτηση νέων μεριδίων στο μετοχικό κεφάλαιο τη Ευρωπαϊκή Τράπεζα για την ανασυγκρότηση και την ανάπτυξη και ευχαριστώ τους Κιώδης για τα χρήσιμα του σχόλια κατά την ανταλλαγή απόψεών μας. Θα προσπαθήσω δε να τα συμπεριλάβω μερικά από αυτά στις τροπολογίες μου. Έχουν υποβληθεί όμως τροπολογίες και από άλλους και άλλες ομάδες και με αυτή την ευκαιρία ζήτησα να διανεμηθεί και μία ορνηθούν ορισμένες προτάσεις συμβιβασμού στους κοιόδης γιατί το πιο εύκολο θα ήταν από το έγγραφο σε αυτό το έγγραφο να βασιστώ για να σε εξηγήσω πού πάμε. Από την αρχή του λοιπόν και παίρνω εδώ υπόψη μου και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Προϋπολογισμών γιατί υπήρχε και ένα θέμα που συνδεόταν με τον προϋπολογισμό θεώρησα ότι έπρεπε και τη δική τους ομοδότηση να την συμπεριλάβουμε. Πρότεινα λοιπόν να δεχτούμε τη γνωμοδότηση 1 που δεν έχει και καμία επίπτωση επάνω στον προϋπολογισμό. Αυτό το λέω στο 3. Μετά προτείνω, όχι στο άρθρο 3, αλλά στην αιτιολογική σκέψη 3. Στην αιτιολογική 6 λέω να συμπεριληφθεί η γνωμοδότηση τρία των προϋπολογισμών. Μα γίνει, υπάρχει θόρυβος και δεν παρακολουθώ λοιπόν. Στην αιτιολογική τα προτείνω τροποποίηση της τροπολογίας μου 9 μετά από πιο πρόσφατες πληροφορίες και προτείνω να λέει σημειώνει ότι η αύξηση είναι για την τριπλή αξιολόγηση, για την τριπλή βαθμολόγηση. Και ότι η αναθεώρηση μετά από την τέταρτη περίοδο που τελειώνει το 2015 μου φάνηκε σωστό να το συνδέσουμε και αυτό με την σωστή περίοδο αξιολόγησης ή αναθεώρησης. Μετά προτείνω να συμπεριλάβουμε και τη γνωμοδότηση 2 των προϋπολογισμών και ο επόμενος συμβιβασμός που προτείνω βασίζεται στην τροπολογία μου 10 και στην τροπολογία 2, 3 και 4 και λέω να λέει ότι ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ΕΤΑ πρέπει να είναι να διασφαλίζει την υποστήριξη νέων αγορών και να μην δίνει δάνεια σε σχέδια για τα οποία υπάρχει χρηματοδότηση με λογικά επιτόκια από άλλες πηγές. Έτσι ώστε να λαμβάνουμε υπόψη μας και τη συνθήκη της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδιαίτερα του άρθρου 21 της. Αυτή είναι η πρότασή μου για τις τροπολογίες εκείνες. Μετά προτείνω να συνδυάσουμε μια από τις τροπολογίες μου και τις τροπολογίες ECR 13 και 14 καθώς και τις 5 και 6 και να λέει λοιπόν η διακυβέρνηση της ΕΤΑ πρέπει να είναι υπόλογη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ετησίως να κάνει αναφορά στην αρμόδιά του Επιτροπή για την προώθηση των στόχων της Ένωσης ιδιαίτερα ως προς τους αναπτυξιακούς στόχους της ε, χιλιετίας, τους στόχους του 2020 και της προοδευτικής κατάργησης της χρήσης άνθρακα καθώς και μεγαλύτερης χρήσης ανανεωσίμων και πιο αποτελεσματικών ενεργειακών πηγών. Έτσι καλύπτω τις τροπολογίες αυτές. Και μετά σε άλλο συμβιβασμό νομίζω ότι μπορώ να συνδυάσω την τροπολογία 11 με την τροπολογία 4 κλούτερ και να λέει να υπάρχει γενικό τεκμήριο γνωστοποίηση των αξιολογήσεων σχεδίων και δικαιούχων τη ΕΤΑ, καθώ και αυστηρότερη έλεγχη για να αποφεύγεται εκ μέρου των δικαιούχων χρήση φορολογικών παραδείσων και το απόρριτο τελεία. Και μου απήντησαν οι σε αυτή την πρόταση λέγοντας ότι πρέπει να ληφθούν υπόψη και η φορολογική παράδειση όπως τους ορίζει ο σαλογική πρόταση μου φαίνεται. Εκτός αν κανείς έχει καμία αντίρρηση. Μετά λέω γενικά να δεχτούμε την τροπολογία 17 αλλά να την αλλάξουμε κάπως για να λέει ότι πρέπει τις πληροφορίες στην ιστοσελίδα να τις κοινοποιεί το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΤΑ σχετικά με τους δικαιούς και τις επιπτώσεις όλων των χρηματοπιστωτικών ενδιάμεσων πράξεων. Μου ζήτησαν όμως μου ζήτησαν όμως να το γράψω λίγο πιο λεπτομερώς, δεν ξέρω αν κανένας πράσινος μπορεί να μας το εξηγήσει. Η τροπολογία 17 είναι η τροπολογία 17 όπου προσθέτω όλα τις τα χρηματοπιστωτικά αποτελέσματα να τα συμπεριλαμβάνει και αυτά στην ιστοσελίδα και τις ενδιάμεσες δραστηριότητες. Μετά προτείνω μια αλλαγμένη διατύπωση της τροπολογίας 13 που να λέει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΤΑ πρέπει να διασφαλίζει, θα συμμορφώνεται προς βασικούς στόχους στρατηγικής 2020 ώστε να ενισχυθεί η συνολική συνοχή των πολιτικών της Ένωσης στον τομέα της εξωτερικής δράσης. και μετά για το 2α νέο που βασίζεται στην 14 και 15 καθώς και στην 20 να λέμε ότι η διοίκηση της ΕΤΑ θα κάνει ετήσιες αναφορές στην αρμόδια Επιτροπή του Κοινοβουλίου για την χρησιμοποίηση των κεφαλαίων της και για τη λήψη μέτρων διαφάνειας ως προς τη χρήση ενδιαμέσων. Τώρα, πώς θα συμβάλλει η ΕΤΑ στην επίτευξη των στόχων και στην συνεργασία με χώρες εκτός Ένωσης με βάση τη συγχρηματοδότηση σχεδίων και προγραμμάτων. Αυτή είναι η συμβιβασμή που προτείνω. Τα σχεδόν όλα υπόψη μου και αναμένω τώρα την ανταπόκριση των σκιωδών. Μερικές αντιδράσεις υπάρχουν ήδη, έχουν υποβληθεί. Ποιος θέλει το λόγο τώρα, ο Ιωάννης Παύλος. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Δεν έχω πολλά σχόλια για τις περισσότερες προτάσεις σας. Απλώς για τη δική μας ομάδα, να πω ότι στην επιλογική σκέψη 10 θα θέλαμε το κείμενο να σταματά στην στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2020. Τρεις γραμμές πριν το τέλο. Αιτιολογική σκέψη 10. Αιτιολογική σκέψη 10 λοιπόν, το κείμενο να σταματά μετά το Ευρω... Ε, η στρατηγική το 2020. Αυτή είναι, αυτό είναι το μόνο μου σχόλιο. Thank you very much. Ευχαριστούμε. Σας ευχαριστώ. Κατά πρώτον, εμείς δεν λάβαμε τις εμβαστικές σας προτάσεις. Δεν μας έχουν αποσταλεί καν. Οπότε και δεν μπορούμε να συζητήσουμε. Επιφυλασσόμεθα λοιπόν να τοποθετηθούμε όταν θα έχουμε διαβάσει τις οπολογίες κυκλοφόρησε ότι κάποιοι θέλουν μια διαδικασία light. Εμείς δεν έχουμε πρόβλημα να συμφωνήσουμε την έκθεσή σας, αλλά τώρα διαπιστώνουμε ότι θα γίνει ευρύτερη συζήτηση, οπότε και επιθυμούμε να γνωμοδοτήσουμε, εφόσον δεν είναι light. Τώρα δεν μπορώ να το κάνω βάσει των προτάσεων σας, τις οποίες ακόμα δεν έχω διαβάσει. Θα δω και τις τροπολογίες των συναδέλφων και θα το μελετήσω. Μας κάνει εντύπωση δεν το εξή. Δεν ξέρω αν η κυρία Λούλινγκ ή κάποιος άλλος συνάδελφος μιλήσουν, κύριος Γκοφέ... η κυρία Λούλινγκ είναι εδώ. Ε, ε λέω ότι μας κάνει εντύπωση το εξή. Έχουν κατατεθεί τροπολογίες, κυριε η κυρια λουλινγκ ειναι εδω λεω οτι μας κανει εντυπωση το εξη εχουν κατατεθει τροπολογιες δυο ας πουμε της κυριας λουλινγκ που θελουν η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης να καταργηθεί και πολύ γρήγορα να ενταχθεί, να απορροφηθεί μάλλον από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Δεν θέλω να προτρέξω, να προεξοφλήσω αυτό που θα πει η κυρία Λούλινγκ, αλλά μια που έχω εγώ το λόγο, καλό θα ήταν, έχει νόημα νομίζω, να πω και τη δική μου γνώμη. Και εγώ πιστεύω ότι Έχουμε τρεις ευρωπαϊκές τράπεζες που πάνω κάτω ε, είναι επενδυτικές. Είναι καλοί οι οργανισμοί, αλλά θα πρέπει εμείς ε, στο Κοινοβούλιο που είμαστε αρμόδιοι να μελετήσουμε κατά πόσο συνεργάζονται αρμονικά και αποτελεσματικά. Και δεν θέλω να σας κρύψω ότι έχω κάποια συμπάθεια για τις απόψεις ε, της κυρίας Λούλιν και του κυρίου Πασκάλ Κοφά στις τροπολογίες τους, γιατί και εγώ έχω παρατηρήσει το εξή έχουμε επικαλύψεις και αναποτελεσματικότητα. Οι τράπεζες τσακώνονται, ανταγωνίζονται μία την άλλη με τρόπο αντιπαραγωγικό. Γιατί θα πρέπει να κάνουμε μια στοχευμένη πολιτική επενδύσεων με το σωστό δυναμικό και δεν μπορούμε σε τελική ανάλυση ε, τρεις τράπεζες να ε, διαγωνίζονται για να πάρει μια τις δουλειές της άλλης, για να το πω έτσι. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Ταυτόχρονα όμως υπάρχει και ακόμα ένα πρόβλημα. Δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε αυτά ad hoc. Βρισκόμαστε σε μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση, σε μια κρίση μέσα σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και τις γειτονικές περιφέρειες. Και η Βόρεια Αφρική βρίσκεται σε δυσμενή θέση αυτή τη στιγμή, οπότε δεν νομίζω να είναι και η βέλτιστη χρονική στιγμή να αρχίσουμε τώρα ε, μια θεσμική αναδιάταξη, αναδιοργάνωση ε, ad hoc. Γιατί οποιαδήποτε νέα διάταξη θεσμών δεσμεύει ενέργεια και δυνάμεις για χρόνια ολόκληρα και αυτό θα είναι εις βάρος της επενδυτικής πολιτικής. Λοιπόν, αυτό είναι μια κλασική σύγκρουση ως προς τους στόχους και εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Αρμόδια Επιτροπή θα πρέπει να δείξουμε φρόνηση. Ποια θα ήταν τώρα μια φρόνιμη συμπεριφορά. Παράδειγμα, δεν ξέρω αν συμφωνείτε κι εσείς ή αν σας προκαλεί χαρά εσάς κυρία Πρόεδρος Συγήτρια ή στους άλλους που έκαναν τις θα μπορούσα να φανταστώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Επιτροπή μας να καλέσει και το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, σύντομα να κάνω μια πρόταση ε, μετά από καθαρή και σε βάθος ανάλυση για την αποτελεσματικότητα της συμπεριφοράς και της δράσης των τραπεζών αυτή τη στιγμή. Και οι δύο να το αναλύσουν αυτό παρακαλώ, και το Συμβούλιο και η Επιτροπή. Και εμείς στη συνέχεια να συνδιαμορφώσουμε τον τρόπο με τον οποίο θα προχωρήσουμε. Αλλά σύντομα ε, σε νέα διάταξη του θεσμικού αυτού αρχιτεκτονήματος. Αυτά όλα πηγαίνουν στην κατεύθυνση των τροπολογιών της κυρίας Λόλινγκ, αλλά είμαστε και εμείς στο τραπέζι. Και η Επιτροπή μας και το Κοινοβούλιο να συνεκτιμά. Γιατί οι τράπεζες έχουν διαφορετικό ιδιοκτησιακό καθεστώς, εξού και διαφορετικά συμφέροντα. Οπότε θα πρέπει στην αξιολόγηση να συμμετέχουμε και εμείς για να δούμε πώς θα λυθεί σωστά αυτό το πράγμα. Και να έχουμε την ε, απόλυτα ακριβή καταγραφή των πραγματικών ε, καταστάσεων και περιστατικών. Αυτά. Αλλά το αφήνω στη συζήτηση. Ακούσουμε και τους συναδέλφους. Yes, I'm, I'm sorry, Udo. Uh, I think what actually... Με Νομίζω ότι ε, αυτό προσπάθησα να προσαφηνήσω με τους υπεύθυνους του γραφείου μου είναι ότι θα είχαν ε, λάβει όλοι σήμερα το πρωί τις τροπολογίες. Αυτομάτως έχουν αποσταλεί όμως ε, στις γραμματείες της ομάδας. Αν κάποιος παραλείψαμε να τις λάβει, λυπούμε ιδιαίτερα. Αλλά θα κάνουμε ό,τι μπορούμε, μπορούμε για να τις λάβετε εγκαίρως τις συμβαστικές προτάσεις. Θα το λάβω υπόψη λοιπόν το στοιχείο αυτό και θα φροντίσω να αποσταλούν όλα με email. Ο Πασκάλ. Ευχαριστώ. Κατά πρώτον, σε ό,τι αφορά εμάς, η καλή συνεργασία που είχαμε και μετά την πρώτη, τον πρώτο γύρο συζητήσεων, η έκθεση άνοιξε και σε κάποια άλλα θέματα και δεν είναι απλώς μια τυπική διαδικασία. Αυτό το θεωρούμε θετικό και εύστοχο, διότι η Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης είναι σημαντική. Η δυνατότητα να αυξήσουμε το μετοχικό μας μερίδιο είναι μια καλή ευκαιρία για να δούμε ζητήματα και διαρθρωτικά και τι αδυναμίες της τράπεζας και έτσι θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το θέμα. Όσο για τις συμβαστικέ σα προτάσει επί τη αρχής μας ικανοποιούν ιδιαίτερω. Όμως πρέπει να πω ότι θα ήταν ιδιαίτερα δυσάρεστο να ακολουθήσουμε την πρόταση του συναδέλφου του Ζαν Πολ, που θαυμάζω κατά τα άλλα ιδιαίτερα ω προ αυτό, διότι αν κατάλαβα καλά πρότεινε να διαγραφεί ακριβώ το τμήμα που αφορά τις δικέ μας τις τη δική μα τροπολογία στην αιτιολογική σκέψη 10 που λέει στη στρατηγική για τη σταδιακή μείωση των συγχρηματοδοτήσεων για κάποια εργοστάσια ενέργειας και τη μεταφορά ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και νέων τεχνολογικών γνώσεων φαίνεται ότι η τράπεζα χρηματοδοτεί ακόμη τέτοιου είδους ε, προγράμματα με δημόσιο χρήμα, κάτι που αντιφάσκει τελείως με τους στόχους για τις κλιματικές αλλαγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει λοιπόν αυτό να ε, επισημαίνεται σαφώς και να υπάρξει σταδιακή μείωση. Αυτό ήδη είναι συμβαστική λύση, διότι εμεί θέλαμε να τεθεί συγκεκριμένη ημερομηνία μέχρι την οποία θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότηση να προτείνει την σταδιακή μείωση. Η ημερομηνία δεν εμφανίζεται καν πλέον στις συμβαστικές προτάσεις. Για σκοπού συμβασμού δεχτήκαμε να γίνει αυτή η διαγραφή. Όμως, προκειμένου να σταματήσει αυτό του είδους ε, η καθάριση και μάλλον αυτού του είδους χρηματοδότηση που αντιφάσκει τελείω με του κλιματικού στόχου τη Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει να αναφέρεται η σταδιακή μείωση. Και όσο για του φορολογικού παραδείσου. Εάν εδώ συμπεριλάβουμε τις, ε, τους συναδέλφους, τις προτάσεις των συναδέλφων για τους φορολογικούς παραδείσους, αυτό ίσως να παρανοηθεί, διότι ο κατάλογος ε, η μαύρη λίστα του ΟΣΑ περιλαμβάνει φορολογικούς παραδείσους οι οποίοι επί της αρχής δεν δέχονται να ανταλλάξουν πληροφορίες μαζί μας. Όμως, το πρόβλημα είναι ότι το να βρεθεί κανείς σε αυτόν τον κατάλογο είναι πολύ εύκολο. Οπότε, ε, οι παρεμηνίε είναι δυνατόν να συμβούν και θα πρέπει εδώ να ακολουθήσουμε τους ορισμούς που είχαμε χρησιμοποιήσει στην έκθεση «Ζολή» ας μείνουμε στα όσα εκεί είχαν εκφραστεί και να μην ξανανοίξει το θέμα εδώ. Είχε γίνει συζήτηση και είχε ψηφιστεί το θέμα αυτό στην Ολομέλεια. Τέλος, είμαι υπέρ τη λύση να γίνει μια σαφής δήλωση για την ανάγκη ευθυγράμμισης των ευρωπαϊκών θεσμών των Ευρωπαϊκών Τραπεζικών Θεσμών. Έτσι κι αλλιώς, στην περίπτωση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων έχουμε πολύ περισσότερο δημοκρατικό πνεύμα από ότι στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης. Για σκοπούς λοιπόν τέτοιας δημοκρατικής ε, μεταχείρισης θα πρέπει να ακολουθήσουμε περισσότερο τις αρχές της τράπεζας αυτής, της ε, Τράπεζας ε, Επενδύσεων, αλλά Υπάρχουν και πολλές επαναλήψεις και επικαλύψεις εδώ. Θα πρέπει λοιπόν να επιδιώξουμε αυτό το στόχο απλοποίησης. Θα πρέπει να αναζητήσουμε και εδώ μια συμβαστική λύση. Uh, thank you. Yes, okay, Mrs. Uh, thank you. Thank you. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κατά πρώτον να σας ευχαριστήσω για τη δουλειά σας. Ευχαριστώ που στηρίξατε και τις τροπολογίες μου. Σε γενικές γραμμές έχουμε ακολουθήσει το πνεύμα των περισσότερων ε, συμβαστικών σας προτάσεων. Απλώς πρέπει να κάνω κάποια σχόλια. Το πρώτο για το ερώτημα του κυρίου Μπούλμαν που το έθεσα πριν από λίγα λεπτά. Καλώς επεσήμανε ότι δεν έχει ακόμα μελετήσει πλήρως ολόκληρο το κείμενο. Ναι, για τις συμβαστικές μιλώ. Απλώς να τονίσω ότι στον κατάλογο των τροπολογιών Η δική μου τροπολογία υπεριθμών 12 νομίζω απαντά στο ερώτημα που κι εσείς σε Αυτό είναι το πρώτο μου σχόλιο. Έπειτα, το δεύτερο απευθύνεται στον κύριο Κοζές. Στο 5C. Τίνω να στηρίξω τη θέση σας και Για μένα ακούγεται λογικό. Για την ΙΕ ε, Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ που δεχτήκατε να γίνει αυτή η προσθήκη βάσει ορισμού του ΩΣΑ διότι αυτό θα κάνει το κείμενο πιο εύληπτο, σαφέστερο. And Τέλος, η συμβαστική F και ο αντίκτυπος των συναλλαγών με οικονομικούς μεσολαβητές εδώ. Χρειάζεται απλώς μια περαιτέρω αποσαφήνιση. Ευχαριστούμε, Άστριτ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχάς να σα πω, ούτε εγώ έχω λάβει τις συμβαστικές σας δεν βρέθηκαν στο γραφείο μου. Εάν τώρα απεστάλησαν, εγώ δεν τις έχω δει. Θα έχουμε το χρόνο να τις συζητήσουμε. Απλώς να πω για την τροπολογία 8, επειδή έγιναν κάποια σχόλια. Εγώ συνεχίζω να είμαι υπέρ της ε, πάυση εργασία τη Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότηση και ανάπτυξη. Εγώ ήμουν υπέρ αυτή τη επιλογή όταν είχαμε κάνει την ε, συζήτηση την τελευταία φορά και οι πράσινοι μάλιστα συμφώνησαν μαζί μου. Μου είχαν πει ότι θα γίνει μια κοινή τροπολογία. Ωραίο είναι αυτό. Αλλά τώρα πρέπει να πω ότι η παράταση της ε, Διάρκεια λειτουργία τη τράπεζας αυτή και προ τη Βόρεια Αφρική. Η παράταση της εντολής φαίνεται να μην βασίζεται σε συγκεκριμένους νομικού. φαίνεται να μην ε, βασίζεται σε συγκεκριμένη νομική βάση, σύμφωνα με το όσα μου είπαν υπεύθυνοι της Επιτροπής ιδίω για τη διεύρυνση τη εντολή προ τη Βόρεια Αφρική. Κάτι που αποφασίστηκε την περασμένη μόλι εβδομάδα. Όπω ξέρετε, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότηση και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ανταγωνίζονται μεταξύ του. Η διεύρυνση λοιπόν τη εντολή τη ε, Τράπεζα ε, Ανασυγκρότηση το επιβεβαιώνει το στοιχείο αυτό, διότι ακριβώ στην νότια ακτή τη Μεσογείου δραστηριοποιείται και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Και πέραν του σκέλου του ανταγωνισμού, που δεν είναι και κάτι το, που το επιδιώκουμε σε κάθε περίπτωση, εφόσον μιλάμε για δημόσιου θεσμού. Εγώ θέλω η εντολή αυτή να εκπληρώνεται, διότι αρχικά Σαφώς θέλαμε να διευκολύνουμε τη μετάβαση, τη δημοκρατική μετάβαση προς την οικονομία αγοράς των χωρών της ε, κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης. Αυτό νομίζω ήταν μια ωραία αποστολή που ανατέθηκε στον κύριο Ταλή. Μεν. Ίσως και να μην ήταν ο μόνος και βασικότερος λόγος, αλλά ήταν σημαντικός. Τέλος πάντων, αφού η αποστολή αυτή εκπληρώθηκε, Νομίζω λογικό θα ήταν να παροτρύνουμε, όπως λέμε και στην τροπολογία αυτή, την συγχώνευση των δύο τραπεζών, δηλαδή την συμπερίληψη της Τράπεζας Ανασυγκρότησης στην Τράπεζα Επενδύσεων. Και θα έλεγα συνάδελφοι να το σκεφτούν όποιος και είναι ο πολιτικός τους προσανατολισμός. Θα εξοικονομήσουμε πολλά μέσα χρηματοοικονομικά μέσα, κάτι που το βρίσκω λογικό σορθό. Είμαι βέβαιη ότι με τον κύριο και με τον κύριο Κονθά μπορούμε να καταλήξουμε σε μια εύστοχη τροπολογία. Και αυτό για να επισφραγιστεί και αυτή η άποψη. Στην τροπολογία μας Άλλωστε, αναφερόμαστε στο ψήφισμα της 22ης Μαρτίου 2009, που καλένε να το θυμόμαστε το ψήφισμα αυτό διαρκώς, διότι σηματοδοτούσε την ε, ορθή οδό που θέλουμε να ακολουθήσουμε. Νομίζω λοιπόν ότι μπορούμε να βρούμε μια τέτοια τροπολογία και βλέπω ότι ο κύριος Μπούλμαν συμφωνεί, συμφωνεί προς τη σύνταξη αυτής της τροπολογίας. Το βρίσκω και λογικό και ε, εύστοχο. Σε κάθε περίπτωση ε, ακούμε επικριτικά σχόλια ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση διασπαθίζει το δημόσιο χρήμα, πόρους, μέσα. Εδώ έχουμε για μια φορά έναν τρόπο να συνενώσουμε, να ομοδοποιήσουμε τις προσπαθίες μας, να γίνουμε πιο λογικοί στην ε, διαχείριση του χρήματος, πιο αποτελεσματικοί. Νομίζω λοιπόν ότι προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει να παροτρύνουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε υπάρχει εδώ ένα μικρό πρόβλημα ότι είναι ευρωπαϊκό θεσμό η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότηση και Ανάπτυξη και έχουμε μόνο το 3%. Αυτό ίσω είναι ένα μικρό πρόβλημα για τι εγχώνε με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Το γνωρίζουμε. Αν είχαμε 100% του μετοχικού κεφαλαίου θα γινόταν. Όμω όταν έχουμε το 3% μόνο, αυτό σημαίνει ότι το υπόλοιπο, το κεφαλαίο βρίσκεται αλλού. Αλλά, άρα όλε οι τροπολογίε έχουν να κάνουν με την ε, διαχείριση αυτή. Ε, έχει ζητήσει όμω το λόγο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν μπόρεσαν ακόμη να με δουν, ε, γιατί ήμουν απασχολημένοι με του τριμερεί διαλόγου. Σφεν, ήθελε προηγουμένω το λόγο. Μια πολύ σύντομη παρατήρηση. Νομίζω ότι πρέπει να έχουμε κατά νου ότι δεν είναι μόνο 3%. Αυτή είναι η επίσημη συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως από πολιτική άποψη μιλάμε για τη συμμετοχή των ευρωπαϊκών κρατών ουσιαστικά, των κρατών μελών. Στηρίζω λοιπόν εδώ την Άστριντ. Έχουμε κάθε νόμιμο δικαίωμα να το συζητούμε το θέμα αυτό, διότι στο κάτω-κάτω τη γραφή μιλάμε για μια de facto τράπεζα των ε, κρατών μελών της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης όπου κατέχουν ένα μέρο του κεφαλαίου. Δεν είναι καθόλου κακό λοιπόν με αυτή την ευκαιρία να συζητήσουμε το όλο θέμα. Στηρίζω πλήρω την Άστρη στα επιχειρήματά τη. Σα ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Απλώ σύντομα να σχολιάσω αυτό που είπε ο κύριο Γκίγκολτ. Αληθεύει ότι όλα τα κράτη-μέλη από κοινού μαζί με του θεσμικού έχουν το 63% στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότηση και Ανάπτυξη. Όμω Πρέπει να θυμόμαστε ότι υπάρχουν και μέτοχοι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και το παρελθόν μας έχει αποδείξει ότι δεν έχουν όλα τα κράτη-μέλη το κοινοτικό συμφέρον κατά όταν συζητούν διάφορα προγράμματα. Θα συνηγορούσα λοιπόν υπέρ της διαφορετικής εξέτασης του κατοχή μετοχικού κεφαλαίου από την Ευρωπαϊκή Ένωση από τα κράτη-μέλη. Μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει το κοινοτικό συμφέρον κατά νου εδώ. Τώρα, για τα όσα συζητήσαμε, ο Επίτροπο γνωρίζει πολύ καλά τον κίνδυνο που προκύπτει από την κατοχή μετοχικού κεφαλαίου και από τα κράτη-μέλη και προσπαθούμε με κάθε δυνατή προσπάθεια να έχουμε αύξηση της αποτελεσματικότητας. Αυτό καλούμε και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και Ανασυγκρότηση και Ανάπτυξη να κάνουν. Να άρουν τι επικαλύψει, να εντείνουν τι προσπάθειέ του προ Ανατολά. Εκεί βέβαια έχουν περιοριστεί ιδιαίτερα επικαλύψει, επειδή δεν είναι ακόμη τόσο ε, ισχυρή εκεί η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ενώ το αντίστροφο συμβαίνει με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότηση. Επίση υπάρχει διαφορετική αντολή για τη μία και την άλλη. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότηση ε, συνεργάζεται με τον ιδιωτικό τομέα ιδιαίτερα στα μεταβατικά στάδια, ενώ η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων με τα μεγαλύτερα επενδυτικά προγράμματα. Για την διεύρυνση στην οποία αναφέρθηκε η κυρία Λούλινγκ, κάτι που πιστεύω διασυνδέεται και με μια σειρά τροπολογιών, θα μας δημιουργήσει το εξή πρόβλημα έχει σχέση με αυτό που είπατε και μόλι τώρα. Δεν είναι ευρωπαϊκό οργανισμό η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότηση και Ανάπτυξη. Δεν είναι υπόλογο μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά στου μετόχου τη, όπου ε, συμπεριλαμβάνονται και η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη τη. Αυτό λοιπόν κάπω περιπλέκει τα πράγματα. Δεν γίνεται να τι ε, αναθέσουμε πολύ σοβαρού κανόνε, πολύ αυστηρού κανόνε υποβολή εκθέσεων. Βεβαίω μπορεί να ζητηθεί να υπάρχει μια λογοδοσία, καθώ οι εκπρόσωποι στην τράπεζα αυτή από την πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση θα προσπαθήσουν να κατευθύνουν και να επηρεάσουν την, το πολιτικό του προσανατολισμό, αλλά και θα πρέπει να λογοδοτούν στο Κοινοβούλιο, να αναφέρονται στο Κοινοβούλιο, αλλά με το 3% δεν μπορούμε να ζητήσουμε κάτι παραπάνω. Και τελευταία μου παρατήρηση ω προ του διαδικαστικού κανόνε. Αυτή η αύξηση του κεφαλαίου έχει περιθώριο εγγραφή ως το τέλος της, ε, του έτους. Έπειτα η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα μπορεί πλέον να έχει περαιτέρω συμμετοχή. Θα πρέπει λοιπόν κάτι να γίνει μέχρι το τέλο τη χρονιά, γιατί αλλιώ το μήνυμα που θα περάσει θα είναι ιδιαίτερα αρνητικό. Πρέπει να στηρίξουμε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανάπτυξη και Ανασυγκρότηση και την ε, διεύρυνσή τη προ την ε, νότια ακτή τη Μεσογείου. Σε αυτέ τι δύσκολε στιγμέ πρέπει να στηριχθεί η τράπεζα αυτή, καθώ η εντολή τη δεν έχει ακόμη πληρωθεί πλήρω. Ούντο, θέλει και... ξανά το λόγο, ναι. Ευχαριστώ, αγαπητοί συνάδελφοι. Ε, νομίζω ότι ακριβώ έτσι είναι ο τρόπο με τον οποίο δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο όπου αμφισβητούνται τα πάντα. Τρέχουμε σε κάθε κράτος μέλος και ρωτάμε πώς μπορούμε να ξεπεράσουμε την κρίση. Ακούμε επικρίσεις για τον προπολογισμό της Ένωσης, ακούμε επικρίσεις από τα κράτη-μέλη για το πόσο είναι ακόμα πρόθυμα να βάλουν το χέρι στη τσέπη για να ανταποκριθούν στις ανάγκες και τις απαιτήσει του κοινοτικού προπολογισμού. Και τώρα κάνουμε εδώ μια συζήτηση που προ τα έξω φαίνεται ότι θα είναι τύχης για τύχα πάντα. Business as usual, συνεχίζουμε, δεν τρέχει τίποτα. Όχι, εγώ είμαι αντίθετο με το πνεύμα που μπήκε τώρα στη συζήτηση στι τελευταίε τοποθετήσει. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Αν έχουμε στοιχεία εμπειρικά ότι είναι τόσο μικρή επικάλυψη, να μα το πείτε. Έχετε αριθμητικά στοιχεία για την Τουρκία, α πούμε, παράδειγμα. Θα με διέφερε. Έχετε αριθμητικά στοιχεία να το στοιχειοθετήσετε αυτό που λέτε, να το τεκμηριώσετε. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων πώ δραστηριοποιείται στην Τουρκία. Ε, η Μπέρντ τι κάνει εκεί, πώ συνεργάζονται και ποια είναι η επικάλυψη. Γιατί με τι συζητήσει που κάνουμε έχουμε αποκομίσει άλλη εντύπωση. Ε, θεωρώ ότι είναι μεγάλη η επικάλυψη και η διπλοδουλειά χωρί να έχω τώρα τα ποσοστά και είναι αναποτελεσματικά. Και το γεγονός ότι έχουν μοιράσει τη δουλειά του θέλει εγώ θα κάνω τις υποδομές, εσύ θα κάνεις τους συμβούλους επιχειρήσεων, ε, δεν είναι σύγχρονος τρόπος λειτουργίας. Και χρειάζεται ε, υπεύθυνη αντιμετώπιση. Κατά τη διάρκεια της κρίσης της ίδιας δεν γίνεται να κάνουμε αλλαγές ε, στη θεσμική αρχιτεκτονική, αυτό το καταλαβαίνω. Αλλά αμέσως μετά και τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να συζητήσουν με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να κάνουν μια ουδέτερη ανάλυση τι πήγε στραβά, ποια είναι τα αναποτελεσματικά στοιχεία και το συντομότερο, όσο πιο γρήγορα μπορούμε, να αναδιαμορφώσουμε την αρχιτεκτονική των δημοσίων τραπεζών μας για να κάνουμε αυτό που περιμένουν από εμά οι ε, ψηφοφόροι μα, να δουλεύουμε αποτελεσματικά. Όταν πάτε εσεί, Πρόεδρε, στην εκλογική σα περιφέρεια, εγώ δεν με ρωτάνε τι πταίει το Συμβούλιο, τα κράτη-μέλη, η Κομισιόν ή το Κοινοβούλιο. Με ρωτάνε Ευρώπη τι κάνει. Κατάφερε να λύσει την κρίση. Αυτό θα πρέπει να τους απαντήσουμε. Και εγώ δεν μπαίνω σε αυτή τη λογική ποιος είναι αυτό το καιρό αρμόδιος. Είναι καλή συζήτηση και ενδιαφέρουσα, αλλά αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να γίνει. Ευχαριστώ. Όπως ξέρετε συνάδελφοι, είμαι εισηγητής εδώ επειδή κανείς άλλος δεν ε, ήθελε να αναλάβει. Φαντάζομαι ότι δεν είναι το πιο διασκεδαστικό λοιπόν από όσο είχαμε να κάνουμε. Σε κάθε περίπτωση. Είμαι ανοιχτή από τις αρχέ για τα θέματα αυτά. Εάν κάποιοι έχουν πρόσθετα σχόλια, θα προσπαθήσουμε να τα λάβουμε υπόψη στις συμβαστικέ προτάσεις, όπου προσπαθήσαμε να καλύψουμε ε, περιπτώσεις όπου Πολλοί είχαν ταυτόχρονα σχόλια. Η τροπολογία της Άστριντ είναι λίγο κατά μέρος, ξεχωριστή. Ε, θα την ψηφίσουμε ούτως ή άλλως, αλλά μετά από τα όσα είπε και η Επιτροπή Άστριντ, ε, ίσως να μην αρέσει ούτε στην Επιτροπή ούτε στο Συμβούλιο, αλλά ούτε και στα κάτι μέλη ένα προς ένα, εάν θες να ακολουθήσεις αυτόν τον προσανατολισμό. Εδώ μιλάμε για το μεταρχικό κεφάλαιο, αλλά από τη μια έχουμε την Ένωση των 100 μελών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και το τι κάνουν ξεχωριστά το καθένα. Μην το ξεχνά αυτό, σε παρακαλώ να το λάβει υπόψη. Επίση, αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε στοιχεία για να μας δείξει κατά πόσο υπάρχουν επικαλύψει ε, και επαναλήψεις, θα ήταν ιδιαίτερα επικοδομητικό να μα τα παρουσιάσει. Σβέν, η Πασκάλ θα θέλαμε και μια πιο συγκεκριμένη πρόταση από εσά, ω προ τον ορισμό που προκύπτει από την έκθεση Ζολή, για να δούμε κατά πόσο μπορεί να γίνει αποδεκτό κάτι τέτοιο. Πάντως, εφόσον ψηφίστηκε η έκθεση αυτή, ε, λογικό ακούγεται. Η μνήμα του ΩΣΑ ήταν μια ιδέα που χρησιμοποιήθηκε συμβαστικά. Βέβαια, καλό είναι να υπάρχει ένα ορισμό στον οποίο πάντα να βασιζόμαστε. Θεωρητικά θα ψηφίσουμε λοιπόν για το θέμα αυτό στι 6 Ιουνίου, οπότε θα ήθελα οι συνάδελφοι να είναι ταχύ στην εξέταση του θέματος και γρήγορα να αποκριθούν στι ε, συμβαστικέ λύσεις που σα προτάθηκαν και ό,τι άλλο θεωρείτε ότι πρέπει να επισημανθεί. Και οι συντονιστές και όσοι υπέβαλαν τροπολογίες καλό θα είναι να τις δουν. Ευχαριστώ λοιπόν όλους τους συναδέλφους. Τώρα περνάμε στο σημείο 5. Κι άλλη έκπληξη. Πάλι κανείς δεν ήθελε να αναλάβει, οπότε εγώ ως πρόεδρος το ανέλαβα. Και αυτό. Νομοδότηση για τις διαδικασίες αφαιρεγγιότητας στο πλαίσιο της νομοθεσίας του εταιρικού δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, νομοθετική, μάλλον έκθεση νομοθετική πρωτοβουλία από την Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων για τι διαδικασίε εφερεγγιότητας, όπως είπα. Αυτά σχετίζονται με τον κανόνα περιθμών 50 και υπάρχει συμφωνία Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων να μην ασχοληθεί με τα ζητήματα τραπεζικής εφερεγγιότητας. Απλώς προσπάθησα να δω ποια θέματα αφορούν τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και θέματα που μας έχουν αποσχολήσει και στο παρελθόν. Όπως θα ξέρετε υπάρχει όριο στους χαρακτήρες. Γι' αυτό λοιπόν στάθηκα στα 7 σημεία, αλλά μπορούμε κάτι ακόμη να προσθέσουμε. Πρώτα απ' όλα φροντίσα να επισημανθεί ότι θα πρέπει η διασυνοριακή ανάκτηση, οι διασυνοριακές διαθήκες ζωής να είναι νομικά εκτελεστές. Εδώ Ξέρουμε από τις συζητήσεις μας για το Solvency 2 ότι όταν μιλάμε για διασυνοριακές περιπτώσεις είναι δύσκολο να γίνουν σωστά αυτά, αλλά είναι κάτι που το επιθυμούμε. Και εδώ μιλάμε για μορφές συνεργασίας διεθνείς που ξεπερνούν τα όρια των τραπεζών. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχουν διαδικασίες εφερεγγιότητας που να επιτρέπουν τον διαχωρισμό των βιώσιμων μονάδων όταν παρέχουν εσωδεί υπηρεσίες όπως συστήματα πληρωμών και άλλους μηχανισμούς που καθορίζονται σε διαθήκε ζωή. Αυτό συνάδει και με τα όσα γίνονται σε διεθνέ επίπεδο για την ε, αντιμετώπιση των κρίσεων. Αλλά και πάλι θα πρέπει όλα αυτά να συμπεριληφθούν στους κανόνες ε, για την αφαιρεγκαιότητα του solvency. Να μην υπάρχει καμία αντίθεση. Επίση, φροντίζω να επισημαίνω ότι οι διαδικασίε αφαιρεγγιότητα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τι μεταφορέ κεφαλαίων. Να μπορεί κανεί δηλαδή να ανακτά στοιχεία του ενεργετικού που έχουν ε, μεταφερθεί για σκοπούς πρακτικούς αυτό θα ήταν χρήσιμο στη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης να ίσχυε ήδη. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι για το διεθνές επίπεδο, αλλά τουλάχιστον σε μια ενιαία αγορά θα μπορούσαμε να το πετύχουμε. Στο σημείο 4. Αναφέρω ότι κάποιες επενδυτικές εταιρείες, ιδίω οι ασφαλιστικές, δεν μπορούν να λύονται αυτή τη στιγμή, ορίζοντας αμέσως πού θα πάνε τα ποσά. Υπάρχουν χρονικά περιθώρια. Βεβαίω, κάποιε επιχειρηματικέ δραστηριότητε μπορούν να μεταφερθούν ή να γίνει αυτό που είναι γνωστό στο Ηνωμένο Βασίλειο Ράνοφ ή κάποιοι άλλοι μηχανισμοί παρόμοιοι. Όμω, θεωρήσα σωστό να λέμε ότι αυτού του είδου οι δραστηριότητε εξετάζονται με ιδιαίτερα χρονικά περιθώρια. Δεν μπορεί να γίνει αυτομάτως η λύση τους, όπως με άλλους ενδεχομένως χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς. Υπάρχει όμως διαφωνία στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τα πόσο εδώ πρέπει να καλύπτονται οι νομικές ε, οντότητες ή ολόκληροι για τι διαδικασίε εφραγκιότητα. Σε κάποιε χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση ολόκληροι όμιλοι παίρνουν στη διαδικασία εφραγκιότητα, ενώ κάποιε άλλε παίρνουν ε, ω βάση τι νομικέ οντότητε. Εδώ συγκεκριμένα, αν και αμφιβάλλω για το κατά πόσον μπορούμε να καταλήξουμε σε ένα απλό συμπέρασμα, εδώ πιστεύω ότι λοιπόν πρέπει να κοιτάξουμε τα ενδεχόμενα αποτελέσματα. Ένα ολόκληρο όμιλο περάσει σε διαδικασία αφαιρεγκαιότητα. Τι διαφέρει από το να μπει μια νομική οντότητα σε αυτή τη διαδικασία. Μπορεί να προκύψουν και άλλα τοπικά προβλήματα ή σε προγράμματα καταθέσεων ή με άλλα εργαλεία που κανείς δεν ήθελε να τα ε, πειράξει μέχρι τότε γιατί δεν, πήγαινε, δεν υπήρχε τίποτα στραβό. Πρέπει λοιπόν να δοθεί έμφαση και σε αυτήν την αλληλεπίδραση εάν θέλουμε να περάσει τη διαδικασία φερεγγιότητα ολόκληρο όμιλο σε μια νομική οντότητά του. Στο 6. Θα πρέπει το εθνικό δίκαιο να μεταχειρίζεται ισότιμα του δανειστέ σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν μιλάμε για την ίδια κατηγορία όμω. Εδώ πρέπει να θυμόμαστε βέβαια και γίνεται με το Equitable Life. Ε, εδώ δεν υπήρχε ίση μεταχείριση για όλου του εμπορευμένου και αυτό πραγματικά ήταν ε, κατά του δικαίου. Αλλά Ακόμη παραμένουν κάποια προβλήματα που δεν τα έχουμε δει. Και το τελευταίο σημείο είναι κάτι που προγραμματιζόταν από καιρό ότι θα πρέπει να υπάρξει ο ειδικό χάρτη για την επίτευξη μια πλήρω εναρμονισμένη διασυνοριακή διαδικασία σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση για την αφαιρεγκαιότητα. Και ότι θα πρέπει να υπάρξει συνένεση και σε διεθνέ επίπεδο. Τουλάχιστον για την περίπτωση μεγάλων χρηματοπιστωτικών ομήλων. Ιδίω ε, για του ε, για τις ενώσεις ομίλων. Εδώ προτίσαμε να αναφερόμαστε σε μεγάλες ενώσεις ομίλων παρά σε μεγάλες ε, ενώσεις χρηματοπιστωτικών ομίλων. Θεωρήσαμε ότι είναι καλύτερο να υπάρχει μια πιο συγκεκριμένη αναφορά. Αυτά είναι τα σημεία στα οποία προφάσισα να σταθώ. Πιστεύω ότι είναι ιδιαίτερα εύστοχα για τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς. Βέβαια θα καλωσορίσω οποιοδήποτε σχόλιο ή συνεισφορά. Ο Ζαν Πολ έφυγε ω συζητητής του ΕΛΚ. Μπούλμαν. Εγώ θα αντικαταστήσω με χαρά το Σαΐντ Αλχαντράουι. Ευχαριστώ πολύ Σάρον για την πρόταση επίσης τη δική σας έκθεση και πάλι έχω την ευχαρίστηση να εκπροσωπώ ως και ο το Σαΐντ και να σας παρουσιάσω τις βασικές μας σκέψεις. Θα ζητήσουμε να υπάρξει ένα σαφές πλαίσιο για τη νομοθεσία σχετικά με την αφαιρεγγιότητα και μάλιστα διασυνοριακή. Ε, κάτι που μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα είναι το εξής. Να υπάρχει και ένα αρμπιτράζ, όχι να έχουμε ένα τουρισμό ε, κατάχρησης ε, νομοθεσίας, να πηγαίνουν οι εταιρείες δηλαδή εκεί που είναι πιο χαραρή νομοθεσία. Όχι. Προοδευτικά να έχουμε στόχο την εναρμόνιση και τους κανόνες εποπτείας και τα διάφορα καθεστώτα. Αυτή είναι η πολιτική μας και αυτή είναι η βάση της. Όλο και περισσότερο βλέπουμε και διαπιστώνουμε ότι αυτό πλήττει και εργαζομένους το θέμα των πτωχεύσεων και θα πρέπει να γίνει πιο εύκολη η διαδικασία της διασυνοριακής εκαθάρισης των επιχειρήσεων, δηλαδή να μην μπλοκάρονται συνέχεια οι διαδικασίες επειδή εκκρεμούν στη δικαιοσύνη να υπάρχουν σαφείς κανόνες και για τη συνοριακή λοιπόν ε, καθάριση και διεκπαιρέωση αυτών των θεμάτων, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για μεγάλες ε, διεθνείς χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις και ιδρύματα, θα πρέπει να βρεθούν σαφείς κανόνες ε, και αξιόπιστοι. Όλα αυτά, κατά την άποψή μας, εντάσσονται σε μια ευρύτερη συζήτηση που είχαμε αρχίσει, θυμάστε, από την έκθεση Φερέιρα για διεθνή και υπερεθνική διαχείριση κρίσεων. Δώσαμε και ολόκληρη έκθεση που θα συνεχίσει την ε, προεργασία της κυρίας Φερέρα. Και θα πρέπει να προσέξουμε οι επιμέρους γνωμοδοτήσεις να συνάδουν με την επιχειρηματολογία που έχουμε πάγια στην Επιτροπή. Ε, αυτά. Ευχαριστώ. Και ο Σαΐντ Ελ θα συνεργαστεί με χαρά μαζί σας. Ευχαριστώ. Σβεν Γκίγκολτ, ζητώ συγγνώμη. Ε, με απασχόλησε εδώ η πρεσβυτέρα. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω ε, πολύ. Στα αγγλικά τώρα. Ε, φαίνεται ότι έχουμε σήμερα κάποιες φαινομενικά ανώδυνες και μικρές εκθέσεις, αλλά με μεγάλη πολιτική σημασία και βαρύτητα. Ε, θα ήθελα να κάνω τα εξή δύο σχόλια. Ε, σχόλια. Σε σχέση με αυτά που είπαμε για τη ε, καθάριση των τραπεζών, θα πρέπει να δούμε ποια είναι η εναρμονισμένη διαδικασία για bailing in και equity swaps. Για την 7η παράγραφό σας, προτείνουμε να οριστεί και να εγκρίνεται ένα οδικό χάρτη για μια πλήρη εναρμόνιση διασυνοριακής εκαθάρισης ε, ιδρυμάτων, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για μεγάλους ομίλους ή ενώσεις ομίλων, με τον ίδιο τρόπο ε, που λέμε ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να βεβαιωθούν ε, ότι το πτωχευτικό τους δίκαιο θα έχει αρκετό περιθώριο για ε, ε, πανευρωπαϊκή εφαρμογή και δράση και ε, να μπορούν να σπάνε οι όμιλοι αν υπάρχουν κάποια υγιή κομμάτια που μπορούν να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους. Άλλος, Ζαν Πολ Γκοζές. Κοίτα, συζητάμε τώρα αυτά τα θέματα της αφαιρεγγιότητας. Θες να πεις τίποτα? Νομίζω ότι θέλεις, έτσι δεν είναι. Είχαμε μια πρώτη συζήτηση για την γνωμοδότησή μου για τις διαδικασίες ε, και ξέρεις ότι εσείς είσαι σκιώδης του ΕΛΚ. Κυρία Πρόεδρε, γνωρίζετε ότι εγώ σας ακολουθώ τυφλά σε όλα τα θέματα με απόλυτη υπακοή και δεν έχω κανένα σχόλιο να κάνω. Ευχαριστώ πολύ. Όπως γνωρίζετε, λέει η Πρόεδρος, το θέμα αυτό το χειρίζομαι από την προηγούμενη θητεία και έχω συνεισφέρει πολύ και στην τότε έκθεση Φεραίρα. Ε, είναι λοιπόν κοινή η αντίληψή μας και χωράει πολύ διεύρυνση και βελτίωση ίσως με τροπολογίες η γνωμοδότηση. Θα καταθέσω και εγώ κάποιες, φαντάζομαι και άλλοι. Η ε, πρόταση τώρα είναι 30 Μαΐου για προθεσμία κατάσταση τροπολογιών. Καλά δεν γίνεται αυτή να παραταθεί. Τι είναι αυτά. Δεν προλαβαίνουμε θεωρητικά να έχετε υπόψη σας ότι 30 Μαΐου είναι. Αλλά θα προτιμούσα να παραταθεί, γιατί φαίνεται ότι χρόνο έχουμε. Μέχρι τις 27 Ιουνίου δεν πρόκειται να ψηφίσουμε. Και η καθελήνα αρμόδια επιτροπή το ψηφίζει στις 19 Σεπτεμβρίου. Το σημαντικό είναι να έχουμε εμεί μια γνωμοδότηση που να μπορέσει να ενταχθεί, να συγχωνευτεί ε, στην έκθεση. Και θα το καταλάβουν φαντάζομαι και θα το σημειώσουν γιατί είναι βάση του άρθρου 50 του κανονισμού. Ωραία, πριν προχωρήσουμε θα ήθελα να καλωσορίσω ένα νέο μέλος, ε, μια αναπληρώτρια από τη Σλοβενία, η κυρία ε, Μάρχα Κρέβ από ε, τη Σλοβενία των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών Κοιτάξτε τι φοβερή δουλειά έχει η πρόεδρος. Τη πέφτουν όλε οι εκθέσει που δεν θέλει κανείς να πάρει. Ερχόμαστε στο σημείο 6. Κοινό φορολογικό καθεστώ το οποίο ισχύει για τι μητρικέ και θητρικέ εταιρείε διαφορετικών κρατών μελών αναδιατύπωση. Μπορεί να είναι πιο συναρπαστικό από ό,τι φαινόταν αρχικά αυτό. Σβέν Γκίγκολτ. Ε, κοιτάξτε να σας πω. Ε, ε είναι και αυτό μια από τις φαινομενικά βαρετές εκθέσεις που όμως τελικά αποδεικνύονται πολύ ενδιαφέρουσες όταν τις εξετάσει κανείς. Στη συνεδρίαση των συντονιστών μας κατηγόρησαν ότι οι μικρές ομάδες εδώ ενδιαφέρονται υπερβολικά μόνο για τα κύρια θέματα και δεν αναλαμβάνουν τα βαρετά. Έτσι αποδεικνύουμε όμως σήμερα ότι δεχόμαστε να αναλάβουμε και τις φαινομενικά βαρετές εκθέσεις για να υπάρχει δικαιότερη κατανομή. Όταν είδα όμως τις λεπτομέρειες διαπίστωσα ότι είναι ενδιαφέρον το θέμα. Γι' αυτό υπάρχει η αναδιατύπωση της οδηγίας για τις μητρικές και θυγατρικές εταιρείες και για την λισαβονοποίησή τους. Δεν μπορούμε βέβαια να συζητήσουμε κάθε λεπτομέρεια της οδηγίας εκείνης γιατί αν και θα χρειαζόταν βέβαια και γι' αυτό θα έλεγα ότι δεν υπάρχει πρόβλημα με τη βασική πρόταση που μας συζητούν να σχολιάσουμε και καθώς αφορά τα φορολογικά δεν ισχύει η συναπόφαση αλλά είναι απλή διαβούλευση για μας. Είναι βέβαια πλήρης έκθεση διότι αν και πρόκειται για ένα απλό τεχνικό θέμα και θα μπορούσε να είχε εξεταστεί και με απλούστερο τρόπο τελικά υπήρξε μια διαμάχη μεταξύ της νομικής υπηρεσίας του Συμβουλίου του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής της νομικές υπηρεσίες και γι' αυτό χρειάστηκε πλήρης έκθεση. Το ενδιαφέρον βέβαια είναι στο αλλαγμένο κείμενο ότι η οδηγία μητρικών θυγατρικών είναι από τους λόγους και το λέω αυτό στην επεξηγηματική έκθεση είναι ένας από τους λόγους για, την λανθασμένη για τον λανθασμένο φορολογικό ανταγωνισμό ενώ θα μπορούσαν πολύ απλούστερα να οδηγηθούν τα φορολογικά έσοδα σε σωστότερους δρόμους και γι' αυτό είναι απαραίτητο να λυθεί το πρόβλημα αυτό. The θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί το CCTV. Είναι όμως ατυχές ότι μέχρι τώρα η Επιτροπή και το Συμβούλιο δεν πρότειναν ουσιαστικέ αλλαγέ τη αρχικής οδηγία, αλλά εμείς στο Κοινοβούλιο τι μπορούμε να κάνουμε. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να τονίσουμε, να θέσουμε το πρόβλημα, γιατί δεν είμαστε σε θέση προς στιγμή να δεχτούμε απώλεια εσόδων από το φορολογικό ανταγωνισμό. Και γι' αυτό η ομάδα μας, η ομάδα μας δέχεται πολλά από τα στοιχεία της αρχικής πρότασης, δηλαδή να εξετάζεται ετήσια η κατάσταση σε μία φορολογική αναφορά που θα κάνει η Κομισιόν κάθε χρόνο. Για να βλέπουμε αν το ισχύον φορολογικό μας σύστημα είναι σωστό, αν υπάρχουν εξαιρέσεις ή φορολογική παράδειση ή διπλή μη φορολόγηση και γενικώ πώς έχει η λεγόμενη φορολογική βιομηχανία ώστε να αποφευχθεί το φαινόμενο που παρατηρείται μια κοινή αγορά να μην έχει κοινούς κανόνες για τη φορολογία και να μπορούν να υπάρχουν φοροδιαφυγές. Στα πλαίσια της έκθεσης αυτής της πρωτοβουλίας έχουν γίνει πολλές ενδιαφέρουσες συζητήσεις αλλά συγκεκριμένα για αυτή την έκθεση τα πράγματα είναι πιο απλά και συστήνουμε στο Συμβούλιο να δεχτεί την λισαβονοποίηση του κειμένου που είναι κάτι με το οποίο συμφωνούμε όλοι και όλες. Σας κατευχαριστούμε. Μάλιστα. Ο Ήβος. Δεν έχω κανένα σκιώδη από το ΕΛΚ που να... Ούντο. Εσύ για τον Λία, εντάξει. Ο Ήβο πρώτος. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Μερικά σύντομα σχόλια που βασίζονται στην επεξηγηματική έκθεση. Υπάρχουν εδώ δύο σημαντικά προβλήματα, θέματα που σχετίζονται με, αυτό το, με αυτή την επεξηγηματική έκθεση. Πρώτον, κάτε με, Το σημαντικότερο είναι πόσο ανεξάρτητοι είναι οι νομοθέτες στον τομέα της φορολογίας και ιδίως της επιχειρησιακής φορολογίας. Όλοι μας φυσικά καταλαβαίνουμε το σημαντικό ρόλο που μπορούν και πρέπει να παίξουν τα εθνικά κοινοβούλια που δικαίω είναι τα αρμοδιότερα για να προετοιμάσουν εθνική νομοθεσία και για την επιχειρησιακή φορολογία. Για μας αυτό είναι το κλειδί μιας κοινοβουλευτικής δημοκρατίας για κάθε κράτος. Αυτό είναι λοιπόν για μένα το σημαντικότερο θέμα που τίθεται. Και το δεύτερο δεν είναι το σημαντικότερο γιατί αυτό είναι ακόμη σημαντικότερο, είναι αν ο φορολογικός ανταγωνισμός μεταξύ των κρατών μελών βλάπτει ή ωφελεί. Εδώ θα είμαι πολύ ανοιχτός. Όλοι μας στην ομάδα μου τουλάχιστον είμαστε υπέρ του ανταγωνισμού και πιστεύουμε ότι ο ανταγωνισμός είναι κάτι το υγιές και επιμένουμε και επί του φορολογικού ανταγωνισμού ως κάτι σημαντικό, υγιές και ωφέλιμο. Ευχαριστώ. Ο Ούντο. Ναι, συνάδελφε Στρέτσεκ, ε, η ομάδα σας ευθύνεται για μια έκθεση από τη δέσμη των 6 ε, που ζητάει μεγαλύτερη τιμωρία και περισσότερες κυρώσεις από τις παρελθόν για τις χώρες που δεν τηρούν το σύμφωνο ε, σταθερότητας και ανάπτυξης. Εκεί οι απόψεις διήστανται και δεν είναι του παρόντος να τις συζητήσουμε. Αλλά ερωτώ, πόσο ευφυές, πόσο συνεπές είναι να λέμε από τη μια ότι στην κρίση και μετά την κρίση στα πλαίσια μιας νέας οικονομικής διακυβέρνησης στην Ευρώπη θέλουμε να τιμωρούμε χειρότερα τις χώρες που δεν φτάνουν στους στόχους για τον προϋπολογισμό και ταυτόχρονα να έχουμε μια φορολογική πολιτική που να την εξηγούμε ε, ε, εν ονόματι του ελεύθερου ανταγωνισμού. Αυτό το αφισβητώ εγώ. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα προχωρήσουμε στην Ευρώπη με τέτοιες ιδέες ανοιχτεί η φορολογική ε, ανταγωνισμή μέχρι να μην μπορεί κανένα κράτος να χρηματοδοτεί αυτά που χρειάζονται από τον προϋπολογισμό τους και όταν δεν το κάνει αυτό να το τιμωρούμε. Ε, τελικά θα επικρατήσει το χάος και θα καταστραφεί η Ευρώπη από αυτή την οικονομικιστική πολιτική και δεν μπορώ να συμφωνήσω με κανένα από τα δύο που είπατε. Εγώ θέλω να συμφωνήσω με τον εισηγητή ε, με τις προειδοποιήσεις τους κατά του φορολογικού dumping. Ε, είναι αρκετές οι μελέτες εμπειρικές, ε, δόξα το Θεό αρκεί να τις διαβάσετε μόνο. Και φαίνεται ότι μπορεί να έχουμε εσωτερική αγορά, αλλά δεν έχουμε κοινή πολιτική και αποφεύγουμε να αναλάβουμε και τις ευθύνες μας. εδώ εκπροσωπώ τον Λία Μνόκ, που είναι ο σκιώδης ηγητής μας, με μεγάλη χαρά τον εκπροσωπώ, και θεωρεί ότι θα πρέπει να κάνουμε περισσότερα από ό,τι προβλέπει η έκθεση. και το λέω και στον κύριο Γκίγκολ, οι σοσιαλιστές και δημοκράτε θέλουμε όχι ένα διατύπωση, αλλά βάθρον διατύπωση ε, ε, και αναγκαστική συζήτηση έτσι, με το ζόρι από την αρχή. Και εκβάθρον να ξαναγραφτεί η έκθεση και θα τα πούμε αυτά και στη συνέχεια. Ωραία λοιπόν. Ε, ο κύριος Μπλουμ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Αν επιτρέπετε να κάνω και εγώ μια-δυο παρατηρήσεις για το θέμα της φορολογίας. Τι είναι ο φόρος. Είναι χρήματα που τα παίρνουμε από τους πολίτες ως πολιτικοί και ουσιαστικά για να δαπανίσουμε για δικά μας, για δικούς μας σκοπούς. Και πραγματικά εδώ μιλάμε για διασπάθηση και σπατάλη. Δεν έχουμε δει πολλά τέτοια φαινόμενα τα τελευταία 15 χρόνια, έτσι σε κάθε περίπτωση στα, στα κράτη-μέλη. Φτάνει πια. Εδώ λοιπόν πιστεύω δεν θα έπρεπε, εάν δεν υπάρχει φορολογικός ανταγωνισμός, πώς θα καταφέρουμε να επιτρέψουμε τη χρηματοδότηση των πολιτικών. Δεν θα υπήρχε καμία βιομηχανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα είχε περάσει όλοι στην Αμερική. Χρειαζόμαστε λοιπόν ανταγωνισμό, αλλά πάνω απ' όλα να πειθαρχήσουμε εμείς οι ίδιοι και να απόσχουμε από τη δική μας την ηλικιότητα. Ζαν ε, Πολ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε να επισημάνω ότι κάποιοι από εμά, όπω ο κύριο Μπλουμ, έχουν μια αίσθηση λίγο σχιζοφρενική. Διότι βρίσκουν του πολιτικού ηλίθιου μένα, αλλά δεν διστάζουν να κάνουν πολιτική καριέρα. Τέλο πάντων, έχω κι εγώ δυο σύντομε παρατηρήσει. Μιλάμε για δημοκρατία. Εγώ, όταν συναντώ του συμπολίτε στην καθημερινότητα, το πρώτο που μου λένε για την Ευρώπη, το δεύτερο τέλο πάντων σχόλιο, είναι δεν καταλαβαίνουμε γιατί στην Ευρώπη δεν υπάρχει ίδια φορολογία σε όλες τις χώρες. Νομίζω ότι και αυτό είναι δημοκρατικό αίτημα. Σε μια ενότητα, ένωση ισχυρή, πρέπει να υπάρχει η μεταχείριση όλων. Ο προσωπικός λοιπόν δεν είναι υπέρ αυτού που ευγενικά αποκαλούμε φορολογικό ανταγωνισμό, αλλά καταλήγει σε κακές αρνητικές καταστάσεις. Και έπειτα, σε ό,τι αφορά την Ευρωζώνη και με την απαραίτητη οικονομική διακυβέρνηση, η φορολογική πειθαρχία είναι μία ανάγκη. Δεν μπορεί να υπάρχει μία ζώνη με νέο νόμισμα. Όσοι είναι κατά του κοινού νομίσματο βεβαίω μπορούν να επιχειρηματολογήσουν κατά. Ε, γι' αυτό βέβαια προφανώ δεν συμμετείχουν κιόλα. Αλλά δεν μπορεί να υπάρχει νομισματική ένωση και όχι φορολογική. Μπορεί να υπάρχει ενθάρρυνση από τη φορολογία ώστε κάποιε επιχειρήσει να παραμείνουν μεν, αλλά δεν μπορεί να γίνεται ανταγωνισμός ε, από μια ευρωπαϊκή χώρα κατά μιας άλλης. Και για όσους λένε ότι είναι κατακράτηση των χρημάτων των πολιτών οι φόροι. Εντάξει, α το δεχτούμε αυτό. Αλλά έναντι φόρου υπάρχουν και κάποιε υπηρεσίε που παρέχονται. Έχουμε κάνει κάποιου υπολογισμούς στη Γαλλία Ιδίω για του Γάλλου που του πλήρωσαν οι πολίτε για να μορφωθούν σε γαλλικέ σχολέ και πάνε και εργάζονται από την άλλη πλευρά τη μάχη. Εδώ, για μια οικογένεια στο Ηνωμένο Βασίλειο, χρειάζεται περίπου τριπλάσιο μισθό από ότι στη Γαλλία για να έχει το ίδιο ποιοτικό επίπεδο σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση, την υγεία και τη στέγαση. Αυτό είναι οικονομική πραγματικότητα να μην την ξεχνάμε, μετά αποφασίζουμε τι θα κάνουμε. Αλλά δεν μπορώ κι εγώ προσωπικά να δέχομαι ότι ο φορολογικό ανταγωνισμός είναι κάτι το θετικό. Υπάρχουν επιτόκια φορολογικά πολύ χαμηλά για τις εταιρείε σε κάποιες ε, χώρες και τα πληρώνουν οι πολίτες. Και αυτό είναι πραγματικό πρόβλημα. Ευχαριστώ, Ζαν Πολ. Το Κένζικτον έχει γίνει πέμπτη μεγαλύτερη γαλλική πόλη ή κάτι τέτοιο. Ότμαρ Κάρας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα συνεχίσω από εκεί που σταμάτησε ο Ζαν Τα άκρα δεν μας βοηθούν να προχωρήσουμε. Και θα πρέπει λίγο να σκεφτούμε τι έχουμε αποφασίσει ως τώρα. Η γεγονό είναι ότι υπάρχει συνθήκη της Λισαβόνας, ξέρετε. Και σε αντίθεση με την προηγούμενη συνθήκη, τον ανταγωνισμό τον έχει κάνει από στόχο μέσο. Λέμε ποια είναι η θέση μας για τον ανταγωνισμό, αλλά δεν είναι και αυτός ο σκοπός. Είναι μέσο ο ανταγωνισμός για να φτάσουμε στους στόχους μας. <laughs> Μετά έχουμε ε, κάνει ε, μοντέλο μας την αηφόρο οικονομία της αγοράς. Και θα πρέπει να είναι ε, το πλαίσιο πιο ισχυρό για να μην πάρουν το πάνω χέρι οι μηχανισμοί της αγοράς. Αυτή η συνθήκη μας δεσμεύει όλους. Επίσης, έχουμε και την πράξη για την ενιαία αγορά, Single Market Act. Από το Μόντι μέχρι το Μπαρνιέ, όλοι για τα φορολογικά ζητούν συντονισμό και κάποια εναρμόνιση τις βάσεις υπολογισμού για τις εταιρείες. Αυτό είναι σημαντικό για την ανάπτυξη και την σταθερότητα και την απασχόληση. Και ένα τρίτο που ακούσαμε προηγουμένως. Το επόμενο βήμα ε, ολοκλήρωσης που είναι οικονομική ενοποίηση δίπλα στην νομισματική το ε, δεύτερο σκέλος επιτέλους να υλοποιηθεί. Και ποιες είναι οι συνέπειες. Γι' αυτό στην έκθεση αυτή ανήκει αυτό το βήμα και στη φορολογική πολιτική για ενίσχυση της εσωτερικής αγοράς και τη δημιουργία και μιας ένωσης ε, κοινωνικής και οικονομικής. Αλλιώς δεν θα έχουμε βγάλει τα διδάγματα που πρέπει από την κρίση. Ευχαριστώ πολύ υποθέτω τα, των φιλελευθέρων θα τα πω εγώ. Συμφωνώ σε γενικές γραμμές ε, με πολλούς από εσά. Ξέρετε τι απόψεις έχω εγώ για το CCCTB ε, και στην περασμένη έκθεση, στην περασμένη θητεία τα είχα πει ε, με κάποιες έτσι παραλλαγές, αλλά μια κοινή φορολογική βάση για μένα είναι ένα σωστό βήμα. Μπορεί να υπάρχουν κάποια προβλήματα. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι θα έχουμε ένα αρμονισμένο φορολογικό συντελεστή. Το CCCTB, θυμίζω, είναι κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιριών. κινδυνεύουν μερικά πράγματα να βρεθούν εκτός ελέγχου μετά από κάποια αποκλιμάκωση που ξεπερνάει το ε, αποδεκτό. Θα πρέπει όμως να αποφύγουμε ε, κάποια ε, διαφυγή ακόμα και αν είναι νόμιμη και το αρμπιτράζ ακόμα και αν υπάρχει, δεν εγγυάται ότι δεν θα φύγει μια εταιρεία για να επωφεληθεί διπλά. Όχι μόνο επειδή θα γλιτώσει τη φορολογία από μια χώρα, αλλά επειδή θα είναι ευνοϊκή και στην άλλη χώρα. Το ξέρω ότι το κοιτάει αυτό ο Σβέν. Είναι πολύ σημαντικό ε, τέτοια παραθυράκια, γιατί παραθυράκια είναι, μπορεί να είναι νόμιμα, αλλά ε, στρεβλώνουν το σύστημα. Αυτά τα παραθυράκια λοιπόν θα προσπαθήσω να τα κλείσω. Προφανώ η κοινή ενοποιημένη βάση φορολογία εταιριών θα το έκανε αυτό. Αλλά δεν σημαίνει απαραίτητο ότι εκεί θα καταλήξουμε. Μπορεί να γίνει σε κάποια κράτη-μέλη και μάλιστα σε θελοντικη βαση βάση τύπου opt-in. Υποθέτω είναι ενδιαφέρον ο τρόπος με τον οποίο σκέφτονται ορισμένε εταιρείε. Αν είχαν μια κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρεών δεν θα μπορούσαν να δρουν όπως δρουν σήμερα. Και η γραφειοκρατία των πολλαπλών συστημάτων νομίζω κοστίζει περισσότερο από ότι η κατάργησή της. Και οι εταιρείε ε, προτιμούν να ιδρύουν θηγατρικές παρά να έχουν διάφορα τέτοια ε, προβλήματα οργανωτικά. Αυτά τα παραθυράκια δεν μ' αρέσουν. Πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρξει ε, όμως ανταγωνισμός ως προς φορολογικούς συντελεστές, όχι ένας ενιαίος συντελεστής για τη φορολόγηση των επιχειρήσεων. Τώρα, στην αναδιατύπωση δεν μπορούμε να κάνουμε και πάρα πολλά πράγματα, απλώς και να κοιτάζουμε, τι χτενίζουμε ε, και κοιτάμε αν μας έχει ξεφύγει τίποτα στρεβλό. Αυτά θα τα ξαναπούμε. Ο κύριος Γκίγκολτ. Δεν ξέρω αν θα είχε νόημα να σας εξηγήσω σύντομα τι στη φόρος. Αλλά έφυγε και όλος ο κύριος Μπλουμ και δεν θα με ακούσει και να τα πω. Κάτι λέει ο κύριος Φέρμπερ δεν ακούγεται χωρίς μικρόφωνο η φορολογία είναι το δικαίωμα του λαού να ψηφίζει για να αποφασίζει πόσο από το εισόδημα θέλουν να δαπανάτε συλλογικά και πόσο ε, ατομικά. Και η διασπάθηση και η σπατάλη γίνεται δυστυχώς και στα δύο επίπεδα, και στον ιδιώτη και στο κράτος. Αλλά και ο ιδιώτης και το κράτος έχει την υποχρέωση να διαχειρίζεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και χρηστή διαχείριση και ε, με βάση κάποιου ηθι... και διεντολογικούς κανόνες. Οπότε η φορολογία δεν είναι κλοπή. Η φορολογία είναι απόφαση να ε, εκτελούμε από κοινού κάποια πράγματα. Και πώς θα καταβάλει το φόρος λοιπόν και με βάση ποιου κανόνες. Εγώ είμαι πολύ μεγάλος υπέρμαχο ε, της ανεξαρτησίας των κοινοβουλίων για να ορίζουν αυτού του κανόνε, αλλά αν είναι πολύ μεγάλη η ολοκλήρωση των αγορών, αυτές οι ανεξάρτητες αποφάσεις δεν μπορούν πλέον να λαμβάνονται σε ε, εθνικό επίπεδο, διότι δεν είναι πια δεδομένη αυτή η ανεξαρτησία. Αν, ας πούμε, υπάρχει ένας φόρος εισοδήματος, θα σηκωθούν να φύγουν τα εισοδήματα. Και αν θέλει κανείς να πάρει σοβαρά ε, το ρόλο του τον ανεξάρτητο, είναι και πιο ευφυές και πιο ανεξάρτητο τελικά να συμμερίζεται κάποιος ε, ε, μια κυριαρχία να είναι στην τρέχουσα αρμοδιότητα. Αυτό είναι καλύτερο παρά να εμένει σε μια υποτιθέμενη εθνική κυριαρχία που πλέον δεν υφίσταται. Και αυτή ε, η κοινωνική ιδεοντολογία οδήγησε στην έννοια και στην αρχή της επικουρικότητας. Επικουρικότητα δεν σημαίνει ότι τα πάντα θα πρέπει να αποφασίζονται στο κατώτατο επίπεδο, αλλά στο κατώτατο το επίπεδο που μπορεί να λαμβάνεται αποτελεσματικά μία απόφαση. Έτσι λοιπόν στη φορολογία πλέον ε, δεν είναι το εθνικό αυτό το επίπεδο. Υπάρχουν λοιπόν πολύ καλοί λόγοι και είδα ότι συμφωνούμε όλοι ε, για μια κοινή ε, ενοποιημένη βάση φορολογίας των εταιριών, αλλά δεν συμφωνώ μαζί σου Σάρων για αυτό που λέγεις για το συντελεστή, το φορολογικό, ότι δεν θα πρέπει να υπάρξει εναρμόνιση αφού είναι τόσο διαφορετικά τα κράτη, να μην είναι διαφορά από το 0 στο 40% όμως από χώρα σε χώρα, γιατί η μηδενική φορολόγηση είναι φορολογικό dumping κατά κάποιο τρόπο. Και καλούμε τις εταιρείες να φύγουν. Όσο κοινή, ενοποιημένη και να είναι η βάση, όσο καλή και να είναι, πάντα χωράει χειραγώγηση. Και αν περάσουμε λοιπόν σε μια κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιριών θα υπάρχει, αν δεν έχουμε κοινό συντελεστή, μεγάλος ανταγωνισμός. Να υπάρχει λοιπόν ένας ελάχιστος φορολογικός συντελεστής ενιαίος και από εκεί και πέρα ένα περιθώριο ε, ελιγμών για τα κράτη-μέλη όπου υπάρχουν πολλά δημόσια αγαθά και αλλού που υπάρχουν λιγότερα. Λοιπόν, αυτό που χρειαζόμαστε δεν είναι πλήρης εναρμόνιση του φορολογικού συντελεστή, αλλά ένα ελάχιστο κατώτατο όριο και ίσως μετά τη συζήτηση αυτή να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε την ψηφοφορία για την έκθεση αυτή, ε, να εκδώσουμε μια μικρή σύντομη δήλωση και να θεωρούμε, να πούμε μάλλον ότι θεωρούμε ε, ότι χρειάζεται να αναδίπωση για να πω και αυτό που είπε ο Ούντο, η οδηγία για τις μητρικές και τις θηγατρικές εταιρείε. Mother-daughter directive, το λένε αυτό στα αγγλικά. Αυτά. Είμαι στη διάθεσή σας, θα με ενδιέφεραν οι απόψει σας. Δυστυχώς ρώτησα τη νομική υπηρεσία και τη γραμματεία, αλλά δεν μπορέσαμε να βρούμε τρόπο να τα λέμε αυτά ε, άμεσα στην έκθεση. Αν έχετε καλύτερες ιδέες έτσι, ως πιο έγκριτη νομομαθής, γιατί εγώ δεν βρήκα τρόπο να μπει αυτό το στοιχείο στη συγκεκριμένη έκθεση. Κρίμα. Κρίμα. Αν έχετε όμως προτάσεις στη διάθεσή σας να τις συζητήσουμε. Ευχαριστώ. Uh, uh, Ευχαριστούμε, Σβέν. Ίσως να πω και εγώ απλώς για να σε διορθώσω ότι μια τροπολογία για τον ε, ελάχιστο φορολογικό. Την έχω. Συγγνώμη, δεν είχα καταλάβει ότι ήσασταν υπέρ του ελάχιστο κοινού συντελεστή. Θα ήθελα μια σαφή δήλωση. Ναι. Άλλαξαν τα πράγματα μετά την κρίση. Η Επιτροπή αυτή είχε ψηφίσει πολλά πριν την ε, κρίση, αλλά δεν θα τα ψήφιζε πλέον. Μάρκος Φέρβερ, τι είπες εσύ και δεν ακούσαμε. Πρόσεχε, εγώ δεν θα έκανα τόσο ε, υπερφύαλες δηλώσεις. Όλοι παιδιά της ιστορίας είμαστε. Anyway, um, and also I, I must say... Μάλιστα. Τα spreads όμως δεν θα φτάσουν ποτέ αυτό το ποσοστό, ακόμη και αν ενοποιήσουμε την ε, βάση. Λοιπόν, ε, τροπολογίες ως τις 20 στις 12 με εξέταση της έκθεσης στις 20 Ιουνίου και ψηφοφορία στην Επιτροπή 21 Ιουνίου. Ολομέλεια στην 1η του Σεπτεμβρίου θα περάσει. Είναι λίγο στενό το χρονοδιάγραμμα, λίγο σφιχτό. Μπορούμε να το παρατείνουμε. Καλό θα ήταν να είχαμε λίγο χρόνο για να κάνουμε και καμιά νομική διερεύνηση του θέματος. Γίνεται να έχουμε μια περαιτέρω διάρκεια για την υποβολή τροπολογιών. Ωραία. Σας ευχαριστούμε. Τώρα, λήξη της συνεδρίασης για το πρωί. Να σας θυμίσω ότι το απόγευμα ξεκινούμε στις 3.30, όχι 3. Αλλά ίσως να μην έπρεπε να σας το πω για να είμαστε όλοι στην ώρα μας. 3.30 πάντως. Και ακριβώς με ψηφοφορίε θα ξεκινήσουμε. Καλό θα ήταν να δείτε τελευταία στιγμή και όλα στο πρόγραμμα, γιατί θα γίνουν αλλαγές και στο κατάλογο ψηφοφοριών. Και παρακαλώ φέρτε τις κάρτες σας και κυρίως ε, των ομάδων. Ευχαριστώ.